Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσουμε τώρα, είμαστε έτοιμοι. Παρακαλώ να καθίστε. Θα ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία ένσταση. Κατά του άρθρου 106 του κανονισμού, ισχυρισμοί υγείας σχετικά με την καφεΐνη. Θα ε, ψηφίσαμε συνολικά για τα εδάφια C, E, I, J και, τεσ, και παραγράφου 4. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Ο κύριος Αφρόντου είναι κατά. Κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τώρα θα ψηφίσουμε το σχέδιο ε, ψηφίσματος. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Ας προχωρήσουμε στην επόμενη ψηφοφορία. για το κείμενο που συμφωνήθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στις άτυπες διαπραγματεύσεις για τα γιατροτεχνολογικά προϊόντα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Θα ε, ψηφίσουμε με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Με συγχωρείτε. Ακόμα ένα. Okay. Ε, ε, the vote is closed. Λύνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται ομοφόνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Now we are going to vote. Τώρα θα ψηφίσουμε. τα διαγνωστικά ιατροτελεφωνικά προϊόντα στην, στο συμβασμό που συμφωνήθηκε μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου ε, στις άτυπες διαπραγματεύσεις. Θα ήθελα να επενθυμίσω μόνον ότι θα περιμένουμε ε, πριν από την, περιμένουμε πριν από την Ολομέλεια δύο δηλώσεις από την Επιτροπή. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσαν όλοι. Κλείνει. Ομοφόνος επίσης. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια. Ας προχωρήσουμε. No flowers for Peter Lise. Okay. Ε, ωραία. Ολοκληρώθηκε. Now we are going to vote. Ψηφίσουμε τώρα. Το θέμα 15, βασική στόχη για την 17η διάσκεψη του ΣΥΤΕΣ των συμβαλόμενων μερών στι ΣΥΤΕΣ. Ερώτηση στην Επιτροπή. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα ε, θα ψηφίσουμε την ερώτηση στο Συμβούλιο. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ολοκληρώσαμε με την ψηφοφορία. Εδώ πέρα θα διακόψουμε και καλούμε τους πάντες να επανέλθουν εδώ ε, για τη συνάντηση με τον κύριο Τίμερμανς στις 5. Ευχαριστώ πολύ.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 Άρα Εντάξει.

Αγαπητοί συνάδελφοι, η ώρα είναι 5 και μπορούμε να ξεκινήσουμε με τη σημαντική συνεδρίαση που έχουμε. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω τον πρώτο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και δεδομένων των πολύ καλών αποτελεσμάτων που έχετε για τα θέματα ε, της βιώσιμης ανάπτυξης θα θέλαμε να ακούσουμε την προσέγγιση της Επιτροπής επί του θέματος και ιδιαίτερα να ακούσουμε για το πρόγραμμα της Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση ε, των στόχων ε, βιώσιμης ανάπτυξης, εξωτερικές και εσωτερικές πολιτικές. Θα θέλαμε να ακούσουμε για την προγραμματισμένη υλοποίηση του προγράμματος κυκλικής οικονομίας. Όπως ξέρετε, ε, η Επιτροπή μας θέλει να παρακολουθεί το πρόγραμμα αυτό τακτικά μέσω ανταλλαγής απόψεων ε, κάθε εξάμεινο μέσα και με τον Αντιπρόεδρο Κατάινεν που επίσης ασχολείται με το θέμα αυτό. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να σας πω ότι μου έχει δοθεί εντολή από το συντονιστή της Επιτροπής ΕΝΒΗ να σας απευθύνω μια επιστολή στην οποία ζητάμε από την Επιτροπή να συντάξει εκθέσεις που θα απευθυνθούν στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης. Την επιστολή αυτή θα τη λάβετε μέσα στις επόμενες ημέρες, αλλά θα ήθελα, μια και είστε σήμερα μαζί μας, να σας το ανακοινώσω για να το γνωρίζετε από σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και σας δίνω το λόγο για την ε, δική σας παρουσίαση και θα ακολουθήσει η συζήτηση με τους συναδέλφους. Θα δώσουμε τη δυνατότητα στους συναδέλφους να κάνουν ερωτήσεις για να μπορέσετε κι εσείς να απαντήσετε. Για τα βασικά σημεία που μας απασχολούν και που έχουμε και στη δική μας ημερήσια διάταξη. Ο κύριος Τίμερμαν, σε ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ για την ε, πρόσκλησή σας. Μετά από την πεσινή μου ε, συνάντηση μαζί σας, όπου ήταν πολύ ευχάριστη η συζήτηση, θα προσπαθήσω στη σημερινή μου παρουσίαση να είμαι πολύ σύντομος. Μπορούμε να συζητήσουμε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και θα αναφέρω το θέμα που εξ αρχής μου ήταν ιδιαίτερα προσφυλές και που θα παραμείνει προτεραιότητα για την πλήρη θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυκλική οικονομία δηλαδή το Δεκέμβριο ψηφίστηκε ένα, μια δέσμη μέτρων και τώρα υλοποιείται το πρόγραμμα δράσης. Και θα σας αναφέρω ως παράδειγμα ότι πριν από δύο εβδομάδες ε, μαζί με τον ε, Κάρλος Μουέδες ε, ξεκινήσαμε τα σχετικά με την υλοποίηση και η Σιμώνα Μποναφέ είναι η συγγήτρια για το σχετικό θέμα στην Επιτροπή σας. Ε, εκ μέρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εμεί είμαστε πρόθυμοι να δώσουμε πλήρη συνεργασία και τεχνικές συμβουλές για να συνδυάσουμε τη φιλοδοξία μας με ξεκάθαρου κανόνες εφαρμογής. Όπως είπα στο Στρασβούργο τον περασμένο μήνα, όταν συζητήσαμε την, το θεματολόγιο των ΗΠΑ για το 2030, είδαμε ότι πρέπει να συνεργαστούμε με πανευρωπαϊκέ λύσει, ε, και όπω είπε και το Ολλανδικό Κοινοβούλιο, αυτή είναι η σωστή λύση και για το περιβάλλον και για τον πλανήτη μας ε, και για το σπίτι μας και για την ευρωπαϊκή οικονομία όμως που απεγνωσμένα χρειάζεται μια νέα όθηση για να υπάρξει επαρκής οικονομική ανάπτυξη που να είναι βιώσιμη ώστε να μας επιτρέπει να χρηματοδοτούμε κοινωνικά συστήματα τα οποία θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικά για την Ευρώπη και που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να βοηθήσουμε και να επενδύσουμε σε τομείς και σε περιοχές γύρω από την Ευρώπη όπου οι προκλήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες λόγω της δημογραφικής εξέλιξης. Άρα τα ζητήματα είναι πολύ περισσότερα και όχι μόνο ε, η οικολογική βιωσιμότητα, είναι και η γεωπολιτική βιωσιμότητα, κάτι το οποίο σχετίζεται απόλυτα με αυτό το θεματολόγιο. Και περνάω σε μια άλλη προτεραιότητα και πρωτοβουλία της Επιτροπής, την βιωσιμότητα. Ε, μέσα στον χρόνο θα ε, παρουσιάσουμε την ε, απόκρισή μας σε θέματα στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Θα παρουσιάσουμε την εξέλιξή μας σε σχέση με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης για να προσδιορίσουμε πού βρίσκεται η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς οι πολιτικές μας μπορούν να συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων που υπάρχουν στο θεματολόγιο 2030. Πέραν ε, του παγκόσμιου χαρακτήρα, το ότι ε, οι στόχοι για την ανάπτυξη είναι στόχοι για ε, τον αναπτυσσόμενο και τον αναπτυγμένο κόσμο, πρέπει από τις κυβερνήσεις να προσδιοριστούν οι στόχοι, αλλά όχι μόνο από τις κυβερνήσεις. Δεν μπορούμε μόνο από την Επιτροπή και από τις κυβερνήσεις να περιμένουμε τον ορισμό των στόχων. Χρειάζεται υποστήριξη και από την κοινωνία των πολιτών και από όλους τους φορείς και από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις περιμένουμε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια καθοριστική συνεισφορά. Η ρύθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θεσπίζουμε την νομοθεσία και πώς ορίζουμε ε, τις ρυθμίσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θέλουμε να συμμετάσχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι για να μπορέσουμε να επιτύχουμε. Και πριν περάσουμε στις ερωτήσεις και απαντήσεις, θα ήθελα να πω δύο λόγια ε, για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Ε, είχαμε αναλάβει δέσμευση πριν από το καλοκαίρι να υποβάλουμε κριτήρια για τον προσδιορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών ε, σε σχέση ε, με την ομοθεσία βιολογικών φυτοφαρμάκων και ο Επίτροπος Ανδριοκάητη σήμερα το πρωί ανακοίνωσε τέτοια κριτήρια που είναι πλήρως ευθυγραμμισμένα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και η προσέγγιση την οποία ακολουθούμε και τα συμπεράσματα τα οποία, στα οποία καταλήγουμε θέτουν ασφαλή κατόφλια και έχουμε αποδώσει ιδιαίτερη σημασία στη σωστή προετοιμασία των εγγράφων τα οποία ανακοινώσαμε σήμερα. Ο Αντιπρόεδρος Κατάινεν και ο Επιτρόπος Αντριουκάητης ε, συνεργάζονται πολύ στενά για να επιτύχουν αυτό το καλό αποτέλεσμα. Ζητήσαμε από τους αρμόδιους φορείς να εξετάσουν ε, τις ε, συγκεκριμένες ε, ουσίες για να μπορέσουμε να οριστικοποιήσουμε τα κριτήρια. Αυτά ήθελα να σας πω και μετά είδα στις ειδήσει σήμερα το απόγευμα ότι διέρευσε ένα έγγραφο. Δεν είναι δική μας πρακτική το να διαραίουμε έγγραφα, αλλά ε, θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια όσον αφορά τις οδηγίες ε, για τα οικοσυστήματα ε, των πτηνών. Είναι πολύ σημαντική η νομοθεσία στους τομείς αυτούς. Είναι πολύ σημαντικές οδηγίες για την προστασία της βιοποικιλότητας. Όλοι γνωρίζουν το δίκτυο Natura 2000 και είχαμε 550.000 ε, απαντήσεις ε, στη διαβούλευση που κάναμε, πάντως πάντω από 500.000 και αυτό δείχνει πόσο σημαντική είναι αυτή η διαβούλευση. Ξέρετε ότι όταν μιλούμε για καλύτερη νομοθεσία, αυτό που πιστεύω εγώ δεν είναι ότι θέλουμε να χαμηλώσουμε τον πύχη, θέλουμε να παραμείνουμε σε πολύ υψηλέ προδιαγραφέ. Και η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν είναι ιδεολογικό το ζήτημα, είναι καθαρά πρακτικό. Και σα το λέω ξεκάθαρα αν κάτι είναι εντάξει, αφήστε το έτσι όπως είναι. Αν μπορούμε να το κάνουμε καλύτερο, να το κάνουμε καλύτερο. Αλλά ε, να μην κάνουμε πράγματα όταν δεν χρειάζεται. Δεν έχουμε ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία. Ε, υπάρχει μια μελέτη σε εξέλιξη και για να ολοκληρώσουμε το έργο μας θα πρέπει ε, να ολοκληρώσουμε το έγγραφο εργασίας το οποίο επεξεργάζεται το προσωπικό της Επιτροπής Θα το δώσουμε στο Κοινοβούλιο πριν από όλους τους άλλους. Ε, εσείς θα είστε οι πρώτοι που θα δείτε την απόφασή μας. Και προτιμώ να ε, συζητήσω με τους συναδέλφους μου στην Επιτροπή, ώστε να γίνει αυτό μαζί με τη συζήτηση που θα ακολουθήσει για το πώς θα προχωρήσουμε παραπέρα. Σας ανακοινώνω λοιπόν ότι εσείς θα είστε οι πρώτοι που θα το μάθετε όταν τελειώσουμε αυτό το έργο και όπως σας ξαναείπα ακολουθώ μια ρεαλιστική προσέγγιση και όχι ιδεολογική προσέγγιση και η άποψή μου είναι ότι αν κάτι δεν είναι σπασμένο δεν χρειάζεται επισκευή. Αυτό ήθελα να πω μετά τη διαρροή από το Euractiv ε, που διέρευσε κάποιες ειδήσεις. Ευχαριστώ πολύ the name of a political group. Ευχαριστώ πολύ. Θα αρχίσουμε τώρα τον πρώτο γύρο των ερωτήσεων από του ΕΛΚ. Πετελίζη από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ, Τζοβάνι. Ευχαριστώ, κύριε Αντιπρόεδρε. Θα ήθελα να αναφέρω τρία σύντομα σχόλια. Αναφέρετε την απόφαση της Επιτροπής για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Εμείς ως ΕΛΚ ε, υπερασπιστήκαμε την Επιτροπή και την αξιολόγηση αντικτύπου, αλλά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, είπε ότι δεν δικαιολογείται καμία καθυστέρηση και επομένω στο μέλλον δεν μπορεί να καθυστερεί τόσο πολύ μια αξιολόγηση αντικτύπου ε, όταν πρέπει να γίνει κάτι πολύ νωρίτερα όταν υπάρχουν ε, κίνδυνοι που πρέπει να αποτρέψουμε ε, ε, για την υγεία, αυτό δεν μπορούμε να το αμελήσουμε. Πρέπει να γνωρίζουμε παραμέτρους όπως η έκθεση και η δόση και διάφορες λεπτομέρειες για το θέμα. Τώρα, όσον αφορά την οδηγία για το fitness check, Έχουμε πει πολλές φορές ότι υπάρχουν θέματα που πρέπει να αλλάξουν, αλλά έχουμε πει ότι μερικές φορές δημιουργούμε περισσότερα προβλήματα από ότι επιλύουμε προβλήματα. Θα ε, σπάμε το κεφάλι μας επί 10 χρόνια για κάποιες τροπολογίες και τελικά ε, θα αρχίσουν να φανάζουν αυτοί οι οποίοι πλήττονται περισσότερο και ε, θα ενοχλούνται και αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι πλήττεται το περιβάλλον και αυτοί τους οποίους θέλουμε να βοηθήσουμε δεν θα έρθουν να μας ευχαριστήσουν και θα έπρεπε να είχαμε βρει κάποια άλλη λύση για τα προβλήματα. Ίσως μερικές οδηγίες ε, δημιουργούν περισσότερο προβλήματα αν πάμε να τις διορθώσουμε από ότι αν τις αφήσουμε ως έχουν. Τέλος, ε, όπως έχουμε πει στο παρελθόν ε, και όπως γνωρίζουμε και από συζητήσεις στην Ολομέλεια για τις διατροφικές αξίες όπου ο ΕΦΣΑ ε, έχει κάνει τις σχετικές ε, δηλώσεις, ε, πρέπει να δούμε ποιες είναι και οι απόψεις της Επιτροπής. Μπορεί κάθε καταναλωτής να ενημερώνεται για το τι υπάρχει σε κάθε είδος διατροφής και πιστεύουμε ότι η γραμμή είναι ότι δεν πρέπει να περιπλέξουμε περισσότερο την κατάσταση με περί τα κατόφλια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, Πίτερ. Ο Ματίας. Ματίας Γκότε, ε, τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν ε, έχει μορφή ακρόαση η συζήτηση. Είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν όλους και έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων. Ε, θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ στο θέμα ε, της ε, οδηγίας REFIT και το θέμα της θέσπισης καλύτερης νομοθεσίας. Είναι πολλά τα προβλήματα τα οποία έχουμε όταν μιλάμε για την υλοποίηση για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε στην πράξη την νομοθεσία. Και για το δίκτυο Natura 2000 έχουμε πει ότι πρέπει να εφαρμοστεί στην πράξη στις συγκεκριμένες περιφέρειες. Υπάρχουν από τη μια μεριά οι αγρότες, από την άλλη μεριά ε, άλλοι ενδιαφερόμενοι και αυτό το οποίο ε, ελπίζουμε είναι ότι ε, αυτό το οποίο πολλοί ελπίζουν είναι ότι δεν θα υλοποιηθεί τίποτα ε, μέχρι να ξεχαστεί το θέμα ή ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Εσείς είπατε ότι θα ακολουθήσετε μια ρεαλιστική και όχι ιδεολογική προσέγγιση. Αυτό το οποίο ε, είναι σημαντικό είναι ότι όταν ε, ε, κάτι αποφασίζεται πρέπει και να υλοποιείται. Αν σε μια διαβούλευση έχουν λάβει μέρος 500.000 πολίτες, περιμένουν ότι κάτι θα προκύψει από αυτή την προσπάθεια. Ξέρουμε ότι ακολουθεί το δημοψήφισμα στη Βρετανία Και ελπίζουμε ότι δεν θα έχει επιπτώσεις σε αυτό το οποίο θέλουμε να επιτύχουμε εμείς με τα ε, νομοθετικά μας κείμενα. Τώρα, Όσον αφορά τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, ε, πρέπει να αναλύσουμε την κατάσταση. Είδαμε και ε, τις απόψεις της Σουηδίας, αλλά ε, ε, πολλοί επιθυμούν ε, μεγαλύτερη ταχύτητα στο πώς χειριζόμαστε τα θέματα για να μην καταλήξουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Για το θέμα της κυκλικής οικονομίας πιστεύω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα τα οποία έχουμε ενώπιόν μας. Είναι ένα πρόγραμμα, ένα πραγματικό πρόγραμμα το οποίο χρειάζεται η Ευρώπη. Έχουμε θέματα τα οποία συζητάμε για την γλυφοσάτη, θέματα τα οποία δημιουργούν μεγαλύτερη απογοήτευση από τίποτα άλλο. Θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη ε, προσπάθεια στο θέμα της κυκλικής οικονομίας για να προχωρήσουμε ε, περισσότερο. Όλοι, ε, όλοι θα υποφεληθούν. Θα υποφεληθούν και οι τοπικές κοινότητες και οι θρησκευτικέ κοινότητες. Ε, νομίζω ότι είναι ένα θέμα στο οποίο μπορούμε να έχουμε ε, ομοφωνία και η κυκλική οικονομία και ο κ. Κατάινεν θα συμφωνήσει. Χρειάζεται λίγο μεγαλύτερη πίεση και η Επιτροπή να μην κουραστεί αλλά να συνεχίσει να υπερασπίζεται αυτό το έργο για την ομάδα μας, για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Η κυκλική οικονομία είναι ένα βασικό θέμα σε αυτή τη θητεία γιατί δημιουργεί δυναμικό για θέσεις απασχόλησης και κινεί την κοινωνία προς τη σωστή κατεύθυνση γιατί σκεφτόμαστε με έναν κυκλικό τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τόμας Μέικορ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την παρουσία σας εδώ στην Επιτροπή μας. Παρακολούθησα με προσοχή τα όσα είπατε σχετικά με το fitness check και την οδηγία Natura. Κύριε Πρόεδρε, μετά από χίλιες μέρες η Επιτροπή δεν γνωρίζει ακόμα τι θα κάνει με αυτή την οδηγία. Ήμουν εισηγητής για, ε, για την αναθεώρηση της οδηγίας για τη βιοπικιλότητα. 86% ε, των βουλευτών ψήφισαν υπέρ της έκθεσης και ζητούσαμε όχι αναθεώρηση των οδηγιών, αλλά πρωτοβουλία για την καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας Natura 2000 ε, και της οδηγίας για τα πτηνά. Μας υποστήριξαν 15 κράτη-μέλη και 500.000 πολίτες οι οποίοι διατύπωσαν τις ανησυχίες τους στα πλαίσια ε, της εκστρατείας alert. Αναρωτιέμαι λοιπόν τι περιμένει ακόμα η Επιτροπή. Δεν μπορούμε να περιμένουμε περισσότερο. Τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνουμε. Και αν έχουμε αυτό το σχέδιο έκθεσης, και την ε, ε, μελέτη αξιολόγηση που υποστηρίζει το fitness check για τις οδηγίες των οικοσυστημάτων και των πτηνών που καλύπτουν 600 σελίδες, επιβεβαιώνεται ότι δεν χρειάζεται να τροποποιηθεί αυτή η οδηγία. Τι αναμένει λοιπόν πλέον η Επιτροπή. Η Ολλανδική Προεδρία θα οργανώσει μια διάσκεψη στο τέλος του μήνα στο Άμστερνταμ και έχουμε ένα έγγραφο εργασίας της Επιτροπής το οποίο θα αναφερθεί για το fitness check. Αυτό το έγγραφο εργασία των υπηρεσιών της Επιτροπής δεν είναι ακόμα έτοιμο. Και αυτό είναι σκανδαλώδες. Προσωπικά αυτό με ενοχλεί πάρα πολύ. Δεν είναι καλή διαχείριση, δεν υπάρχει διαφάνεια και δεν είναι δημοκρατική διαδικασία. Πράγματι η επιθυμία μας είναι να πετάξετε από το παράθυρο ε, την μόνη εμπιστοσύνη που μπορεί ακόμα να έχουν, την τελευταία, το τελευταίο ίχνος εμπιστοσύνη που μπορεί να έχουν οι πολίτες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι απαράδεκτο. Η Επιτροπή μας λέει ότι φταίει η κρίση των προσφύγων. Αλλά επειδή έχουμε μια προσφυγική κρίση, αυτό δεν είναι δικαιολογία. Γνωρίζω ότι είναι μεγάλη πρόκληση, είναι τιτάνιο το έργο, αλλά η βιοπικιλότητα είναι ένα πρόβλημα και εδώ δεν μπορούμε να χάσουμε χρόνο. Ε, δεν σας κατηγορώ προσωπικά, αλλά αυτή η καθυστέρηση είναι απαράδεκτη. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτή την κατάσταση. Γιατί περιμένει ακόμα η Επιτροπή, ποιος είναι ο πραγματικός λόγος αυτής της καθυστέρησης. Δουλέψαμε σκληρά για αυτές τις οδηγίες και θέλουμε ε, να υπονομεύσουμε τη δουλειά που έκαναν μερικοί. Ποιος θέλει να υπονομεύσει τη δουλειά τους. Υπάρχουν ε, ε, ομοσπονδίες μηχάνων που βρίσκονται πίσω από αυτές τις ενέργειες. Προφανώς εκλήθησαν οι σύνδεσμοι βιομηχάνων για να μας συζητήσουν το θέμα. Γιατί δεν έχουμε ένα έγγραφο εργασία από τις υπηρεσίες της Επιτροπής για να συζητηθεί το Άμστερνταμ. Πότε να μας δώσετε κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Γκερμπράντι. ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να απευθύνω ένα θερμό καλώ όρισα μα στον ε, Επίτροπο Φραν Τίμερμαν. Συζητούμε κάτι που ίσω ε, μακροπρόθεσμα θα είναι το σημαντικότερο ερωτήμα του χαρτοφυλακίου του. Μπορεί να μην ε, παίρνει την πολιτική προσοχή που το αρμόζει, αλλά σε 10-15 χρόνια θα το αντιληφθούν όλοι ότι ήταν πραγματικά το σημαντικότερο κομμάτι του χαρτοφυλακίου σε σχέση με το όσα είπε για το μά ο κύριο δεμές Μάκερ για την οργή για τα οικοσυστήματα, δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπε, όμως θέλω να τονίσω δύο πρόσθετα στοιχεία. Πρώτον, πόσο χρόνο, ε, πόσος χρόνος χρειάστηκε η Κομισιόν. Αυτό δημιουργεί τεράστια ασάφεια. Τι θα συμβεί δηλαδή με τη μελλοντική νομοθεσία Natura. Θα μετριαστεί ε, το περιεχόμενό της, γιατί αν υπάρχει αυτό το άνοιγμα, τα κράτη-μέλη και τα κοινοβούλια ε, θα ε, αποφασίσουν. Κανείς δεν ξέρει λοιπόν τι πρόκειται να συμβεί. Και αν δείτε όλες τις αναλύσεις για τις πολιτικές στην Ευρώπη, σε αφορά το Natura, είναι ίσως από τα πιο επιτυχημένα νομοθετήματα του τρέχοντος κοινοτικού κεκτημένου. Ένα πρόβλημα υπάρχει μόνο, η εφαρμογή από τα κράτη-μέλη. Αν όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίσει ε, να δαπανά τόσο χρόνο για τη διαδικασία REFIT, τελικά θα ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν την εφαρμογή. Ή θα σημαίνει αυτό ότι θα περιμένουν και αυτά περισσότερο χρόνο πριν εφαρμόσουν τις διατάξεις. Μάλλον το δεύτερο θα συμβεί αυτό φοβάμαι τουλάχιστον. Δεύτερον, ενδιάμεση αναθεώρηση βιοπικιλότητας. Όλοι συζητούμε και λέμε πόσο σημαντική είναι η φύση εν γέννη και υπάρχουν πολλές μελέτες που δείχνουν και από οικονομική πλευρά ότι η βιοπικιλότητα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σε παγκόσμιο επίπεδο η απόλυτη τη βιοπικιλότητα υπολογίζεται ότι κοστίζει 3% σε ανάπτυξη του ΑΕΠΑ ετησίω. Τρία χρόνια, 3% ε, κάθε χρόνο χάνουμε. Άρα, όταν ο Οργανισμό Περιβάλλοντο, ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντο, δημοσίευσε την κατάσταση για το Natura πέρυσι τον Απρίλιο, πάνω από χρόνο δηλαδή, συγκάλεσε πολλές έκτακτες συνδριάσεις κομισιών, επειδή προσπαθούμε όλα περνοσμένα να πετύχουμε την οικονομική ανάκαψη και εδώ φάνηκε ότι η απώλεια της βιοπικιλότητας δεν έχει ανακοπεί σε καμία περίπτωση, που σημαίνει ότι η η μελλοντική απώλεια θα επηρεάσει και την οικονομική ανάκαμψη. Επειδή λοιπόν δεν έχουν γίνει πολλά μέχρι τώρα, βλέπουμε τα πορίσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την αναθεώρηση στρατηγικής για τη βιοπικιλότητα και βλέπουμε να έχουμε το ίδιο καταστροφικό συμπέρασμα ε, που συνήγαγε και η Επιτροπή, ο Οργανισμός Περιβάλλοντος, δηλαδή δεν θα ε, πετύχουμε τους στόχους και δεν θα ανακοπεί αυτή η απώλεια της βιοπικιλότητας. Ούτε έχουμε ανακτήσει την απώλεια που έχουμε ήδη. Εγώ περιμένω λοιπόν εναγωνίως τις προτάσεις της Κομισιόν για το πώς θα φύγουμε από αυτό το αρνητικό μονοπάτι και πώς θα πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει το 2020, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα έχουμε τα ίδια ε, συμπεράσματα με το 2010, ότι δηλαδή δυστυχώς δεν πετυχαίνουμε τους στόχους. Τέλος, κύριε Πρόεδρε, να πω και δύο λόγια για την κυκλική οικονομία. Η γλώσσα μας είναι μια χαρά και εσείς χρησιμοποίησατε πολύ ωραία γλώσσα πέρυσι, αλλά εδώ δεν είναι οικονομικό το θεματολόγιο, είναι, δεν είναι περιβαλλοντικό, είναι οικονομικό συγγνώμη το θεματολόγιο και μιλάμε για την μελλοντική οικονομική ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως ε, δεν φαίνεται ότι ε, τα έργα τα αποκρίνονται ε, εντελώς στα λόγια πολλά και πολλές είναι οι διαδικασίες για την κυκλική οικονομία που όμως επιβραδύνονται. Στην διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξάμεινου δεν έχει μείνει τίποτα για την ε, κυκλική οικονομία. Ε, το eco-design το είχατε υποσχεθεί για το 2015 και αυτό επιβραδύνθηκε και έχει αναβληθεί. Επαόριστον από ό,τι γνωρίζουμε. Διαφωτίστε μας λοιπόν σας παρακαλώ σε σχέση με τις πολιτικές προτεραιότητες της κυκλικής οικονομίας. Είναι ακόμη μόνο μια ένα προτεραιότητα ή πάνω-πάνω τέλο πάνω στι προτεραιότητε, ή έχουμε να κάνουμε μόνο με λόγια και όχι με έργα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ΚΟΕ. Κύρια Κονέτσνα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας ε, σήμερα εδώ και μακάρι να μπορείτε να μας επισκέπτεστε πιο συχνά στην Επιτροπή μας τουλάχιστον μια φορά το χρόνο θα θέλαμε να σας έχουμε εδώ. Θα μπορούσαμε να επωφεληθούμε από την επίσκεψη αυτή, γιατί είστε υπεύθυνο για πολλά θέματα για τα οποία είμαστε και εμείς αρμόδιοι και ελπίζουμε ότι θα σας βλέπουμε συχνότερα και δεν θα χρειάζεται να περνάει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως ήδη ανέφεραν οι προλελήσαντες, θα ήθελα και εγώ να μιλήσω για τις ε, οδηγίες για τα πτηνά και τα οικοσυστήματα και για το κατά πόσο η Επιτροπή επιθυμεί να τις ε, ανανεώσει. Μέχρι τώρα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι και ήταν πολύ δυσάρεστη έκπληξη η δήλωση του εκπροσώπου τύπου της Επιτροπής. έχουν τόσα πολλά πράγματα να κάνουν σε σχέση με την κρίση του προσφυγικού που δεν προλαβαίνουν να κάνουν κάτι άλλο. Ήδη δεν τα πήγε πολύ καλά η Επιτροπή σε αυτά τα θέματα. Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιούμε σαν πρόφαση και για άλλους τομείς. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Επιτροπής ότι ε, δεν θα κάνουμε τίποτα και απλώς θα περιμένουμε να λυθεί το προσφυγικό για να κάνουμε κάτι άλλο. Ε, ε, εκτός από την οδηγία για τα πτηνά και το οικοσύστημα υπάρχει και το θέμα για τα απόβλητα και η αξιολόγηση αποβλήτων για τον Natura 2000. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να δούμε κατά πόσο έχουν εφαρμοστεί όλα αυτά στα κράτη-μέλη. Γιατί νομίζω ότι αποφασίζουμε νέες οδηγίες, νέες διατάξεις και τα κράτη-μέλη δεν ε, ακολουθούν. Και θα ήθελα να ε, κάνω ένα σχόλιο και για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες που είναι θέμα που όλους μας απασχολεί. Ε, δεν είναι σωστή η στάση του Επιτρόπου Αντριοκάητης, διότι φαίνεται να ε, μην δίνει καθόλου σημασία στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Θέλουμε οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα θεσμικά όργανα, αλλά όταν η ίδια η Επιτροπή δεν σέβεται τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, πώς θα γίνει αυτό. Θα ήθελα λοιπόν η Επιτροπή να ασχοληθεί με το θέμα. Πολύ για τους πράσινους τώρα, η κυρία Οούκεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. θα παρακαλούσα τον Επίτροπο να ακούει τα Ολλανδικά, επειδή η μετάφραση είναι πολύ καλή στα Ολλανδικά. Φυσικά, είπαν αυτά που επρόκειτο να πω εγώ σχετικά με το refit το οποίο δεν χρησιμοποιείται, το οποίο λυσμονούμε. Θα έλεγα λοιπόν στους συναδέλφους, δεν είναι σωστό αυτό απέναντι στον Επίτροπο είπε ότι δεν πρέπει κανείς να αλλάξει κάτι που είναι καλό. Είναι πολύ σαφές το μήνυμά του. Εάν οι οδηγίες είναι καλές, όπως ακούμε, αυτό λέμε στις εκθέσεις μας, δεν αλλάζει κανείς κάτι που είναι καλό. Και τελικά η Επιτροπή χρησιμοποιεί τις λέξεις που χρησιμοποίησαμε εμείς παλιότερα. Νομίζω ότι είναι σαφές. Πρέπει να συγχαρούμε τον Επίτροπο. είναι κανείς πιο χαρούμενος όταν βλέπει κάποιον να μετανοεί. Πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τον Επίτροπο οι συνάδελφοι ρωτούν τι πρέπει να γίνει, τι είναι το σημαντικό. Ε, ο Επίτροπος να ακούει τις θαυμάσεις συμβουλές που θα του δώσουμε. Το σημαντικό εδώ είναι όπως είπαμε η βιοκυπηχηλότητα, όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά για, την, για το κλίμα. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Η σωστή βιοπικιλότητα. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ελπίζουμε να δραστηριοποιηθεί η Επιτροπή και να κάνει το καταδύναμη. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχει φωτιά. Δεν πρέπει όλοι να καούμε σε αυτή τη φωτιά, κυρίως στα πλαίσια της νομοθεσίας, ε, η οποία είναι αρεστή στους πολίτες μας. Δεν πρέπει να είμαστε αδύναμοι, διότι τότε οι πολίτες θα δουν ότι είμαστε αδύναμοι. Πρέπει να δείξουμε ότι τα πράγματα πάνε καλά, ότι είναι κάτι που μας αρέσει, να το ενισχύσουμε, να το αποδεχθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος ερωτήσεων από τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Δίνω λοιπόν το λόγο στον πρώτο αντιπρόεδρο κύριο Τίμας για το πρώτο γύρο απαντήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω τους βουλευτές για τα σχόλια και τις ερωτήσεις τους. Σε ό,τι αφορά τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, φυσικά αυτό που έγινε σήμερα ήταν μια απόπειρα να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει πλήρη συμμόρφωση με τι αποφάσει του δικαστηρίου και αν είναι σωστέ οι πληροφορίες μου, αύριο θα το συζητήσετε το θέμα με τον Επίτροπο Άντριου Κάιτης, ο οποίος θα μπορέσει να σας δώσει και όλα τα στοιχεία της σημερινή απόφαση. Και νομίζω ότι περιμένει με ανυπομονησία αυτή την ανταλλαγή απόψεων με τους ευρωβουλευτές σε ό,τι αφορά τα πτηνά και τα οικοσυστήματα. Ξέρετε, κάποιες φορές ε, σε εσωτερικό επίπεδο τα πράγματα ε, καθυστερούν περισσότερο από όσο θα ήθελα. Έτσι είναι η ζωή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, κάποιες φορές εμείς περιμένουμε να αγωνίω στον ορισμό εισηγητών από μέρους σας και αργεί πολύ κάποιες φορές. Άρα αυτά συμβαίνουν σε όλα τα θεσμικά όργανα. Στην προκειμένη περίπτωση ε, το δουλεύουμε, το προσπαθούμε. Σας παρουσίασα τη δική μου γενική προσέγγιση. Και στα Δανέζικα άκουσα ε, πολύ καλά και με έντονο τρόπο ε, τι πιστεύετε. Σίγουρα μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα. Πώς, αυτό θέλω να ξέρω, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να εφαρμόσουν ε, τις σχετικές διατάξεις στα κράτη-μέλη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διαφυλάσσοντας την βιοπικιλότητα της χλωρίδας και πανίδας. Για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό που έχουμε δει, το είπε και ο και Μπράντι νομίζω, είναι ότι συχνά το πρόβλημα έγκυται στην εφαρμογή της νομοθεσίας όταν αυτή μεταφέρεται στο εθνικό δίκαιο. Εκεί πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βοηθήσει τα κρατημέλη για να αποφευχθεί η ασάφεια και ούτω καθεξής. Αφού τα λέμε όμως εδώ ειλικρινά και ανοιχτά, να πω και κάτι ακόμη. Δεν λαμβάνω πάντοτε τα ίδια μηνύματα από τις ίδιες πολιτικές ομάδες, τα ίδια πολιτικά κόμματα. Πολλές φορές λαμβάνω πολύ έντονα συναισθηματικά μηνύματα. Ο κύριος Ντεμεσμάκερ τα είπε εδώ, όμως κάποιοι από τους ε, ίδιους ε, από τους συναδέλφους του στο ECR, στην ίδια πολιτική ομάδα, έχουν εντελώς ε, διαμετρικά αντίθετες απόψεις και βασίζονται στους ίδιους πολίτες λέγοντας ότι αυτοί δεν θέλουν να το κτλ. κτλ. Επομένως, το να επικαλείται κανείς τους πολίτες δεν πάντοτε καλύτερη προσέγγιση. Εγώ όμως, τι να σας πω, εγώ βασίζομαι σε ξύσμα του κοινοβουλίου, πράγματι. Σας είπα ποια είναι η δική μας γραμμή, η δική μου γραμμή. Μην με κατηγορείτε όμως ότι ψεύδομαι, γιατί αυτό κύριε Δεμεσμάκερ δεν θα το ε, λάβω υπόψη ελαφρά την καρδία, δεν το δέχομαι από κανέναν. Άρα, αν με κατηγορείτε για ψεύτη, αποδείξτε το. Εγώ δεν σας λέω ψέματα, σας τα λέω πολύ απλά, είμαι πάντοτε ειλικρινής και ανοιχτός και σας λέω ότι αυτά παίρνουν χρόνο, λυπούμε γι' αυτό, θα ήθελα και εγώ να είχαμε προχωρήσει πιο γρήγορα, απλά όμως παίρνει χρόνο. Τι να κάνουμε. Εγώ θέλω ε, να σας παρουσιάσω ε, το ολοκληρωμένο προϊόν, όταν έχει ολοκληρωθεί όχι μόνο την ανάλυση της δημόσιας διαβούλευσης δηλαδή, αλλά και την αντίδραση της Κομισιόν. Θα έχουμε ένα υπηρεσιακό έγγραφο εργασία. και θα σας παρουσιάσουμε και τα μηνύματα που πρέπει να δώσουμε προς τα έξω. Αυτή η συνάντηση σήμερα νομίζω ότι είναι πράγματι ένα χερό μήνυμα. Μην με παρεξηγείτε λοιπόν. Νομίζω ότι υπάρχει στο Κοινοβούλιο πολύ μεγάλη πλειοψηφία που μου δίνει πολύ σαφές μήνυμα. Ο εκπρόσωπος του ΕΛΚ ξεκίνησε ακριβώς με αυτό έδωσε αυτό το μήνυμα και το εκτιμώ ιδιαίτερο. Γιατί και αυτό ήταν ειλικρινή και είπε ποιε είναι οι του για το που βαδίζουμε και προ ποια κατεύθυνση κινούμαστε. Θα με βοηθήσει αυτό όταν χρειαστεί να λάβουμε αποφάσεις εσωτερικό επίπεδο στην Κομισιόν. Μην επιτίθεται λοιπόν ένας στον άλλο. Καλύτερα να συνεργαστούμε να είμαστε στην ίδια πλευρά όταν ε, τραβάμε το σκηνή, όχι ο ένας από τη μία και ο από την άλλη. Και εσείς και εμείς λοιπόν, από τα θεσμικά όργανα τα οποία υπηρετεί ο καθένας μας, να μελετήσουμε καλά τα πράγματα, ώστε να είναι σαφείς οι αποφάσεις που θα πάρουμε στο τέλος. Τώρα, ο κύριος Λίζε είπε για τα διατροφικά προφίλ, που δεν εγκρίθηκαν ποτέ. Και τώρα κάνουμε μια αξιολόγηση για να δούμε τι πρέπει να γίνει. Και νομίζω ότι του χρόνου αναμένονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής. Στρέφομαι τώρα στην κυκλική οικονομία. Θέλω να επαναλάβω για μια ακόμη φορά ότι πρέπει την κυκλική οικονομία να την συμπεριλάβουμε σε όλες τις δράσεις μας. Δηλαδή, αν δούμε τις δυνατότητες της ενέργειας ψηφιακής αγοράς, την ε, ανάπτυξη και την δημιουργία μιας ενεργειακής ένωσης, βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ό,τι κάνουμε επίσης ε, στον τομέα των υποδομών κτλ. Το ΕΦΣΙ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, έχει πολύ ενδιαφέρουσε συνιστώσει στο ταμείο αυτό. Αν δούμε επίσης πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα διαρθρωτικά ταμεία. Α προσπαθήσουμε όλα αυτά ε, να τα συμπεριλάβουμε σε μια προσέγγιση βιώσιμης οικονομίας, κυκλική οικονομία ω βιώσιμη οικονομία. Και τα κράτη-μέλη θα λάβουν τις συστάσεις μας πρέπει να τονίσω κάτι που είπε ο κύριος Γκρότε και ο κύριος Γκερμπράντι. Θέλουμε να έχουμε μια πραγματική αλλαγή παραδείγματο στην οικονομία μας. Και σίγουρα είναι πολύ μακρόπνο και φιλόδοξο αυτό το όραμα. Αν δείτε τις νέες επενδύσεις μέσω του ΕΦΣΥ και υπάρχουν και πραγματικοί στόχοι μάλλον το πόσο διαφορετικά. Το γεγονό ότι στην αγορά υπάρχει τόσο πολύ ενδιαφέρον σημαίνει ότι Κάποιες φορές ε, οι αγορές, οι επιχειρήσεις, οι διάφοροι κλάδοι της βιομηχανία σκέφτονται ίσως περισσότερο στρατηγικά από ότι εμείς. Και εμείς πρέπει να τους βοηθήσουμε να οδηγεύσουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Γνωρίζουμε που βρισκόμαστε προς την οικονομία και που πρέπει να πάμε. Δεν είναι τεχνική η πρόκληση, ούτε επιστημονική. Δεν είναι ούτε καν ε, δημοσιονομική, οικονομική. Είναι μια πρόκληση που έχει να κάνει με την πολιτική βούληση και τι ρυθμίσει, του κανονισμού. Γι' αυτό θεωρούμε ότι η καλύτερη νομοθεσία, οι καλύτερες ρυθμίσεις θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο νομοθετούμε και να συμπεριλάβουμε πολύ περισσότερο ΜΚΟ, άλλους συμπληκωμένους φορείς και θα φτάσουμε έτσι σε ένα σημείο που η νομοθεσία θα είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκε τη μετάβαση προ την κυκλική οικονομία. Τα Green Deal, οι πράσινες συμφωνίες ε, εντάσσονται σε αυτή την προσέγγιση με τον Κάρλος Μοέδας ε, που προκύξαμε αυτό το διαγωνισμό, ε, αυτό, σε αυτό αποσκοπούσαμε και στην Ολλανδία βλέπουμε κάποια project τις τελευταίες ημέρες που εν μέρει χρηματοδοτούνται από το ΕΦΡΟ και αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα πρόκληση για εμάς στην Κομισιόν αλλά φαντάζομαι και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι αυτό αφορά όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης εντάσσεται στην γενική προσέγγιση SDGs, στους αθλητικούς στόχους, στους ε, στόχους, αλλά πολλά θα πρέπει να γίνουν και σε εθνικό επίπεδο. Και πάμε όμως και στο τοπικό επίπεδο, γιατί, για παράδειγμα, δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει πολιτική για τα απόβλητα που θα είναι βιώσιμη, αν δεν συμμετέχουν εκεί οι τοπικές αρχές. Άρα η πρόκληση είναι πρόκληση διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα. Και ρύθμιση επομένου. Νομοθεσία. Συμφωνώ λοιπόν απόλυτα με τον κύριο Χερμπράντη. Άκουσα πολύ προσεκτικά όσα υπόθηκαν για τη βιοπικιλότητα. Και συμφωνώ. Ε, άρα θα προσπαθήσω, ο συνάδελφος που μου έθεσε κάποια ζητήματα, να προσπαθήσω να εφαρμόσω αυτά που μου ζήτησε. Δεν ξέρω μέχρι που μπορώ να φτάσω. Θα επανέλθω όμως, γιατί επίστην ότι είναι κατεπίγουσα κατάσταση λόγω της απειλής που δέχεται η βιοπικιλότητα. Σας άκουσα λοιπόν τώρα τι μπορώ να κάνω δεν ξέρω, αλλά τα σημειώνω όλα αυτά και ίσως επανέλθω και εδώ κύριε Πρόεδρε στην Επιτροπή σας άπαξ και έχω ε, εντοπίσει τι μπορούμε να κάνουμε για να επιταχύνουμε τα πράγματα και να βελτιώσουμε την κατάσταση. Νομίζω, ναι, τους ενδοκρινικούς διαταράκτες απάντησα. Νομίζω τις περισσότερες ερωτήσεις έχω απαντήσει κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα μπορούμε να περάσουμε στο δεύτερο γύρο των ερωτήσεων από τα μέλη. Ο κύριος Μπέλετ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, δικαίως υπογραμμίσατε τη σημασία της κυκλικής οικονομίας, την πολιτική, οικολογική και γεωπολιτική σημασία που έχει η κυκλική οικονομία σε τοπικό επίπεδο τα μισά απορρίμματα πηγαίνουν σε χώρους υγειονομικής ταφής στις κοινότητες. Γι' αυτό αυτός ο στόχος είναι ο πιο προφανής, ίσως και ο πιο απλός να αντιμετωπιστεί, δηλαδή να μην γίνεται υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, αλλά να γίνει προσπάθεια για ε, αναδημιουργία, ανακύκλωση Φυσικά πρέπει και να στοχεύει πιο ψηλά, μεσοπρόθεσμα, και ο στόχος θα είναι να αποφεύγονται τα απορρίμματα, τα απόβλητα, τα οποία περιέχουν και πρώτες ύλε. αλλά πρέπει τα προσεχή χρόνια ε, να αποφεύγουμε να ενισχύουμε επιφυακά μοντέλα που δεν είναι τα κατάλληλα, διότι έτσι θα ενθαρρύνουμε τη δημιουργία ε, ενέργειας, στην παραγωγή ενέργειας με βάση τα απόβλητα και τελικά ε, θα βρεθούμε παγιδευμένοι μέσα σε επενδύσεις που κάνουμε σήμερα. Γι' αυτό πιστεύω ότι ήδη από σήμερα πρέπει να στοχεύουμε πιο υψηλά τα απόβλητα. Δεν θα πρέπει να είναι απόβλητα, αλλά θα πρέπει να τα δούμε σαν πρώτες Και η ενέργεια ίσως είναι μια ψευδής λύση, θα πρέπει να ανακυκλώσουμε τα απόβλητα και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ίσως δεν είναι η σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Ο, ο Αντιπρόεδρος κύριος Πρότσο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καλωσορίσατε κύριε Αντιπρόεδρε. Finally. Δεν θέλω να επαναλάβω πράγματα που έχουν λεχθεί, αλλά νομίζω ότι αρκετέ παρανοήσει έχουν προκύψει τους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο χρόνο μεταξύ τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα σα δώσω κάποια παραδείγματα. Είπατε και συμφωνώ ότι δεν θέλετε ε, κάτι που δεν είναι σπασμένο να προσπαθήσετε να το επισκευάσετε. Άρα γιατί ακούμε και συζητάμε θέματα σχετικά με ε, οδηγίες που δεν έχουν κανένα πρόβλημα ε, γιατί να θέλει η Επιτροπή να κουμπίσει οδηγίες όπως ε, για τα πτηνά, για τα οικοσυστήματα. Φαντάζομαι ότι ε, ε, και εσείς θα έχετε λάβει πολλές διαμαρτυρίες, ε, όπως έχω λάβει και εγώ, γιατί πολλές διαμαρτυρίες προέρχονται και από την ίδια τη χώρα σας. και για τα χωροκατακτητικά είδη το ίδιο ισχύει. Ε, γιατί η Επιτροπή, ε, η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος προτείνει κάτι για ε, τομείς που χρειάζονται λιγότερο από οποιοδήποτε άλλο τομέα κάποια αλλαγή. Αποφασίζει η Επιτροπή να ακολουθήσει μια πορεία με πολιτική χρειά και όχι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες το ίδιο. Δεν σας κατηγορώ ότι ψεύδεστε, κάθε άλλο. Ίσως όμως να έχετε εσφαλμένη ενημέρωση για τον ορισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών. Δεν είναι ίδιος με τον ορισμό της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Ο ορισμός της Επιτροπής είναι πιο αδύναμος. Υπάρχουν λοιπόν αρκετά επικίνδυνα σημεία. Θέλω να παραμείνω με θετικό πνεύμα και θέλω να σας ρωτήσω πώς νομίζετε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε καλύτερα σε θέματα που είναι πολύπλοκα. Πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερη επικοινωνία μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Δεν το γνωρίζω γιατί υπάρχει αυτή η νέα οριζόντια δομή. Μερικές φορές μας λένε ρωτήστε τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής, αλλά δεν ξέρουμε ποιον αντιπρόεδρο της Επιτροπής να ρωτήσουμε. Ε, τι συμβουλή λοιπόν έχετε να μας δώσετε, πώς θα μπορούσαμε να επικοινωνούμε καλύτερα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί μερικέ φορέ μα διαφεύγει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε που ήρθατε σήμερα. Κατά σύμπτωση, πριν από λίγες εβδομάδες άρχισα να διαβάζω την έκθεση για την Ευρωπαϊκή Διαβούλευση για το θέμα της ε, βελτίωσης καταλληλότητας του κανονιστικού πλαισίου και μου έκανε μεγάλη εντύπωση το νούμερο. 500.000 τόσοι πολίτες απάντησαν. Από αυτό το μισό εκατομμύριο απαντήσεων που λάβατε, οι 520.000 προέκυψαν από μια αυτόματη πλατφόρμα, όπου απαντά κανείς δύο-τρεις ερωτήσεις με αυτόματο τρόπο. Μόνο το 3% όλων των απαντήσεων 16.850 συγκεκριμένα έδωσαν λεπτομέρειες σε σχέση με τις ερωτήσεις ε, που τέθηκαν στη διαβούλευση. Αυτό το μοντέλο διαβούλευσης με ενοχλεί. Γιατί και για την TTIP ίδιο μοντέλο διαβούλευσης ακολουθήθηκε. Και προσπαθεί, προσπαθούν κάποιοι να μονοπολίσουν την ε, δημόσια συζήτηση. Αυτό το είδος λοιπόν τεχνολογίας με ενοχλεί ως πρώην δημοσιογράφο και με ενοχλεί πάρα πολύ διότι εν μέρη χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και από εσά. Δεν είναι ηθικά αποδεκτό και θα ήθελα την απάντησή σας από αυτού. Ευχαριστώ. Σε ποια συγκεκριμένη ερώτηση θέλετε απάντηση, γιατί άκουσα τη δήλωσή σας, αλλά ερώτηση δεν άκουσα, λέει ο Επίτροπος. Ο κύριος Κάνατε μια δημόσια διαβούλευση η οποία στρεβλώνεται λόγω των αυτοματοποιημένων απαντήσεων. Δεν πρόκειται για συζήτηση μεταξύ πολιτών. Είναι μια ε, αυτοματοποιημένη διαδικασία και οι απαντήσεις βγαίνουν μέσα από ένα αυτοματοποιημένο σύστημα. Πώς κρίνεται αυτό το σύστημα. Ευχαριστώ πολύ. Με συγχωρείτε που άλλαξα τη σειρά. Κανένα πρόβλημα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον Τίμερμανς σχετικά με την αυξανόμενη προσφυγή στην επιτροπολογία από αυτή την επιτροπή, δηλαδή και το κοινοβούλιο. Ε, προσπαθούμε να περιορίσουμε την επιτροπολογία και ο ρόλος τη Επιτροπής είναι πολύ σαφής. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να γνωμοδοτήσουν και η Επιτροπή μπορεί να υιοθετήσει τις εφαρμοστικές πράξεις. Αυτά που βλέπουμε με τα, τους οργανισμούς, τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και δεν ξέρω ότι πιστεύει η πλειοψηφία εδώ είναι ότι δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα. Και γνωρίζω ότι η Επιτροπή προσπάθησε να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα να βοηθήσει στο μέθοδο του δυνατού χωρίς επιτυχία. Γι' αυτό υπήρξε μια δυσλειτουργία εδώ. Και βλέπουμε όλο και περισσότερο και σε άλλους τομείς πολλές αντιρρήσεις και ορισμένε ε, οδηγούν τις επιτυχίες στην Ολομέλεια, αλλά όλες ε, έχουν πολιτικά κίνητρα. Ε, μετά από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η Επιτροπή οφείλει να τηρήσει τις νομικές υποχρεώσεις και επίσης ε, υπάρχει και απόφαση του συνηγόρου πολίτη για την κακοδιοίκηση και τις καθυστερήσεις. Και να ρωτιέμαι εσείς ε, κατά πόσον, για να εξασφαλίσετε καλύτερη νομοθεσία, πώς προτείνετε να γίνουν αλλαγές προκειμένου ε, να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Thank you very much. Now, Mr. Eck. Eck. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε Τίμερμανς, θα ήθελα να μιλήσω για το θέμα της κατασπατάλησης ε, μέτρων διατροφής σε σχέση με την κυκλική οικονομία. Η πρόσφατα δημοσιευθήσα έκθεση του 2016 δηλώνει ότι δεν έχουν γίνει ε, αρκετά για να καταπολεμήσουμε την σπατάλη στα ε, είδη διατροφής, ε, παρότι υπάρχει ε, ε, σημαντικό πρόβλημα στις χώρες οι οποίες πλήττονται από έλλειψη ειδών διατροφής θα μπορούσε λοιπόν μια τροποποίηση της γεωργικής πολιτικής να βοηθήσει σε αυτόν τον τομέα για να επιτύχουμε τους στόχους που έχουν τεθεί γιατί ο τρόπο με τον οποίο τρεφόμεθα εμεί στην Ευρώπη και ο τρόπο με τον οποίο παράγουμε μέσα διατροφή έχει ε, άμεσε ε, επιπτώσεις στην παγκόσμια ασφάλεια των μέσων διατροφής και ε, επίπτωση στις χώρες του τρίτου κόσμου που υποφέρουν από έλλειψη μέσων διατροφής. Σε σχέση λοιπόν με την κατασπατάληση μέσων διατροφής, θα ήθελα να σας ρωτήσω κύριε Αντιπρόεδρε αν η Επιτροπή θα κάνει συγκεκριμένες προτάσεις στο πλαίσιο της καλύτερης νομοθεσίας για να ε, μεταρρυθμίσει την γεωργική πολιτική και να επιτύχει τους στόχους του 2030 και αν θα έχει η Επιτροπή το θάρρος να αντιμετωπίσει το μοντέλο της υπερπαραγωγής με τρόπο οικολογικά βιώσιμο, ώστε το μοντέλο που θα έχουμε να αποφεύγει τη σπατάλη ειδών διατροφής στην Ευρώπη. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε ε, που είσαστε κοντά μας σήμερα και ελπίζουμε να μην είναι η τελευταία φορά. Θα ήθελα να θίξω τρία θέματα. Τα δύο πρώτα αφορούν ε, την προσευχική εργασία που έχει κάνει η προηγούμενη Επιτροπή σχετικά με τον Επιτροπό Σκοτώσνικα. Ένα είναι ένα έγγραφο ε, που αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη που αποτελεί τη βάση για την συμμετοχή ε, των πολιτών στη δικασία λήψης αποφάσεων και συμβάλλει ε, σε βιώσιμες οικονομίες και κοινωνίες και είναι απαραίτητη για την εφαρμογή της σύμβασης που προβλέπει κατάλληλη πρόσβαση στη δικαιοσύνη των ε, πολιτών. Το θέμα είναι ότι η Νέα Επιτροπή σχεδιάζει να επανέλθει σε αυτό το θέμα το οποίο είχε ξεχαστεί κατά κάποιο τρόπο από τη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντα η Νέα Επιτροπή και πότε μπορούμε να αναμένουμε κάποια πρωτοβουλία από τη Νέα Επιτροπή σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Το δεύτερο θέμα είναι παρόμοια φύση πάλι. Ε, η Επιτροπή Ποτάτσνικ είχε προετοιμάσει ένα έγγραφο της για τις, ε, ε, τους ελέγχους που γίνονται στα θέματα περιβάλλοντος. Όπως γνωρίζουμε, οι επιθεωρήσεις του περιβάλλοντος που γίνονται ε, είναι πολύ σημαντικές για την εφαρμογή ε, της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρώπης και κυρίως ως επειδή οι επιθεωρήσεις περιβάλλοντος είναι ευθύνη των κρατών μελών. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ κρατών μελών και μερικές φορές αυτές οι διαφορές δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στην εφαρμογή ε, της κοινοτικής νομοθεσίας. Μπορούμε να περιμένουμε ότι μετά από δύο χρόνια η Επιτροπή θα επανέλθει σε αυτές τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις. Και το τελευταίο θέμα αφορά την οδηγία για τα οικοσυστήματα και τα πτηνά που αναφέρθηκε επανειλημμένος. Πιστεύω ότι ήδη πολλά ελέγχθησαν και εγώ θα ήθελα ένα ερώτημα να θέσω. Μπορείτε να πείτε ποια θα είναι η προθεσμία την οποία η μελέτη σχετικά με το REFIT θα είναι έτοιμη. Μπορούμε να περιμένουμε ότι η Επιτροπή θα δρομολογήσει το σχέδιο δράσης, υλοποίησης της οδηγίας οικοσυστημάτων και πτηνών. Διότι αυτά είναι τα προβλήματα με τις οδηγίες. Ευχαριστώ. Κυρία Κώστιγκερ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής. Και εγώ θα ήθελα να μιλήσω για το θέμα της ε, καλύτερης νομοθεσίας σε σχέση με ε, το Natura 2000. Υπάρχουν τόσα πολλά παραδείγματα από τα κράτη-μέλη όπου βλέπουμε ότι ε, θα είχε νόημα να έχουμε μια πιο ευέλικτη στάση για την προστασία ε, της φύσης ε, νομίζω ότι ε, υπάρχουν σημεία που θα έπρεπε να αλλάξουν και αν μπορούμε να έχουμε θετικές επιπτώσεις θα μπορούσε η οδηγία να προσαρμοστεί και από τη δική μου περιφέρεια θα μπορούσα να σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει μια μεγάλη πρωτοβουλία πολιτών που έθεσαν ως στόχο να επαναφέρουν στην περιοχή μας ένα είδος πέστροφας που υπήρχε πριν από πολλά χρόνια και μην γελάτε, μπορεί να ακούγεται αστείο, αλλά είναι σημαντικό ότι ε, υπάρχει η νομοθεσία και ε, όλοι λένε ότι οι Βρυξέλλες φταίνε που δεν μπορούμε ε, να το κάνουμε γιατί ορίζεται το απόθεμα των αλευμάτων κατά τέτοιο τρόπο. Είναι τέτοια πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία οι πολίτες ε, αντιμετωπίζουν. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε ε, να ακολουθήσουμε ένα συγκεκριμένο μέτρο ή ότι φταίνε οι μονοκαλλιέργειες, αλλά υπάρχουν κάποια προβλήματα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη. Άλλο ένα θέμα είναι τα δικαιώματα των ε, ιδιοκτητών. ξεχνάμε μερικές φορές ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν εκεί και δουλεύουν εκεί και θέλουν ε, να διατηρήσουν τον τόπο τους ε, με τρόπο βιώσιμο. Και πολλές φορές οι άνθρωποι απογοητεύονται λόγω της νομοθεσίας που ισχύει. Μπορώ να σας δώσω παραδείγματα όπου με μονομένοι ε, αγρότες ε, οι οποίοι ζουν από ε, την ξυλία την οποία κόβουν. Δεν είναι μεγάλες μονάδες ξυλίας, αλλά από αυτό τον τομέα ε, ζουν και απογοητεύονται και στρέφονται κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, γιατί ε, θα μπορούσαμε να δώσουμε σε αυτούς τους απλούς πολίτες, σε αυτούς τους αγρότες μία θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να ακουστεί και η δική του η φωνή. Προσπάθησα να σας δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα για να σας δείξω ότι για όλους μας είναι σημαντικό να βελτιωθεί η κατάσταση. Ξέρω ότι έχετε πολλά να κάνετε και πρέπει να ασχοληθείτε και με αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Euh, θα πω ότι σας ευχαριστήσω για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Εξετίμησα ιδιαίτερα τα όσα είπατε σχετικά με την κυκλική οικονομία που είναι ένα από τα μεγαλύτερα διακυβεύματα όχι μόνο για να καταπολεμήσουμε τις κλιματικές αλλαγές αλλά και για να καταπολεμήσουμε την ανεργία παντού στην Ευρώπη τα προσεχή χρόνια. Αύριο στις 14 θα συναντήσουμε τον κύριο Αντρουκετή, τον Επίτροπο Υγείας, που παρουσίασε στο Κολέγιο των Επιτρόπων σήμερα το πρωί το νομοθετικό πακέτο για τους ε, ενδοκρινικούς διαταράκτες. Τώρα δύο θέματα. Εξ όσων γνωρίζω, ο κατάλογος των ενδοκρινικών διαταρακτών περιλαμβάνονται στα παραρτήματα που παρουσιάστηκαν σήμερα το πρωί από τον Επίτροπο στο Κολέγιο των Επιτρόπων. Αλλά σε αυτή την αίθουσα, στο κύκλιο ή στον πανόροφο, πολλές φορές ε, αναφέρατε ότι είχατε δεσμευθεί επανειλημμένα για να επιτρέψετε πριν από το καλοκαίρι τη δημοσίευση των ενδοκρινικών διαταρακτών, του καταλόγου δηλαδή. Και το θέμα είναι, μπορείτε να επιβεβαιώσετε αυτά τα οποία λέω, εφόσον δεν υπάρχει ακόμα ο κατάλογος. Επίσης, ε, είναι ευκαιρία να δείξουμε ορισμένα θέματα που δεν είναι τόσο επίκαιρα, ε, που δεν αφορούν ίσως του διαταράκτες ή την κυκλική οικονομία, αλλά ένα θέμα το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Είναι εκείνο της διαφάνειας και άλλωστε και σας ενδιαφέρει. Δηλαδή, ποιες είναι οι σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των λόμπιστ, δηλαδή για να υπάρχει διαφάνεια. Εσείς θέλετε να αλλάξετε ε, όλο το θέμα της διαφάνειας. Όπως ξέρετε, η ε, συνήγορος του Ευρωπαίου Πολίτη λέει ότι μερικές φορές δεν υπάρχει διαφάνεια στις σχέσεις μεταξύ ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καπνοβιομηχανίας και ε, συναντήσεις με τους λόμπιστε και δεν έχουν γίνει σεβαστές οι αποφάσεις τους εκτός της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Προστασίας Καταναλωτών. Από τη στιγμή όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση επικυρώνει και υπογράφει ε, την ε, σύμβαση του, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας για την καταπολέμηση του, του καπνίσματος, πρέπει να εξασφαλίζεται και διαφάνεια και αυτό αναφέρεται άλλωστε τις συστάσεις της, όπου ζητείται προληπτικά να δημοσιεύει τα πρακτικά όλων των συναντήσεων με τους καπνοβιομηχάνους. Στην περίπτωση λοιπόν ε, της μεταρρύθμισης ε, ε, του φακέλου της διαφάνειας, θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας. Ευχαριστώ κύριο Σουίτεμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ κύριε Αντιπρόεδρε. Έχω μια ερώτηση σε ό,τι αφορά τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τη διαδικασία διοδότησης. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια διέξοδα ε, από θεσμικές με το γλυφοζάτ ε, τελευταία. Δεν θα πρέπει ταυτόχρονα ε, να βασίζεστε σε επιστημονικά δεδομένα αλλά και με βάση μια δημοκρατική διαδικασία. Τα κράτη-μέλη που πρέπει να συναποφασίσουν όμως φαίνεται ότι η απρόθυμα ή ανίκανα είναι να καταλήξουν σε συμφωνία. Γι' αυτό και σας έχουν ξαναστείλει τον μπαλάκι. Το Συμβούλιο δεν αναλαμβάνει τις ευθύνε του, δεν τοποθετείται και επομένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή που θα πρέπει από μόνη της να αποφασίσει και τελικά είναι αυτή που ε, κατηγορείται και για όλα τα κακά των αποφάσεων που λαμβάνει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν πώς βλέπει αυτή την κατάσταση και τι σκοπεύει να κάνει για να λύσει αυτή, αυτά τα θεσμικά διέξοδα που προκύπτουν συνεχώς. Και επόμενο ερώτημα, τα απορρίμματα από τρόφιμα. Τι κάνετε ε, στο πλαίσιο του δέσμης μέτρων ε, για την διαχείριση των αποβλήτων με αυτά τα αποβλήτα συγκεκριμένα και την κυκλική οικονομία. Κυρία Πύρικ, Σράιερ Πύρικ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πρέπει να σας πω ότι όταν έρχονται ομάδες επισκεπτών από τις κάτω χώρες και τους ε, μιλώ για την κυκλική οικονομία και το ΕΦΣΥ, το βλέπουν ε, ιδιαίτερα θετικά. Οι πολίτες αλλά και η βιομηχανία στις κάτω χώρες είναι θετικά διακείμενη. Θα έλεγα μάλιστα ότι είναι και αυτό που σε ενδιαφέρει περισσότερο. Βέβαια υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Για παράδειγμα, γνωρίζουν, οι δύο νέοι που κάποιοι είναι και πίσω στην αίθουσα, ε, τι θα πει κυκλική οικονομία. Μιλάμε για πολύτιμε θέσει εργασία. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε περισσότερο. Και τώρα έρχομαι σε δύο-τρία συγκεκριμένα σημεία. Μιλάμε για τον τομέα των αποβλήτων. Αν δείτε τι γίνεται στι κάτω χώρε και με την κυκλική οικονομία, μόνο το 1% των αποβλήτων ε, πηγαίνει σε χιτά. Αλλά αν δείτε τι γίνεται, για παράδειγμα, στην Πορτογαλία ή αλλού, υπάρχουν μεν καλές ιδέες, αλλά υπάρχουν και πολλά εμπόδια. Θα μπορούσαν ε, κάποιο είδος απόλυτα να χρησιμοποιηθούν στην ε, οικοδομή, ως δομικό υλικό. Είπατε ότι θέλετε να βρείτε λύσεις και χαίρομαι γι' αυτό. Είπε και η αυστριακή συνάδελφος ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Και ο κύριος ε, Ντέμες Μάκερ είπε ότι υπάρχουν ε, πολλά email που παίρνουμε από τις οργανώσεις προστασίας ε, περιβάλλοντος κτλ. Εγώ είμαι και μέλος Επιτροπής Αλίας. Και πρέπει να σας πω ότι θα μπορούσα να τα μετρήσω σε 3-4 εκατομμύρια αυτά τα email που λαμβάνω και που λένε ότι κάτι πρέπει να γίνει για την προστασία της φύσης. Άκουσα και τον κύριο Χερμπράντη. Και δεν είναι μόνο οι αγρότες, όλοι οι Ολλανδοί πολίτες αλλά και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό. Να σας δώσω κάποια άλλα παραδείγματα. Δεν μπορούμε πλέον να κάνουμε ποδήλατο επειδή υπάρχουν κάποιε προστατευόμενες περιοχές. Δεν μπορούμε επίσης να κατασκευάσουμε κάποιες ε, οδούς ε, πλακόστρωτα, παραδείγματος χάρη γιατί πρέπει να προστατεύσουμε τις νυχτερίδες και ούτω καθεξής. Στην Ολλανδία έχουμε πρόβλημα. Δεν μπορούμε επίσης να φροντίσουμε για τη διατήρηση κάποιων ε, περιοχών ε, όπου κάνουν τη φωλιά τους, τα πτηνά κτλ. Υπάρχουν, ξέρετε, και οικογένειες που επί εκατονταετίες ε, οικογένεια, γενιά, μια γενιά μετά την άλλη ε, εκμεταλλεύονταν τη γη και δεν μπορούν πλέον να το κάνουν. Υπάρχει ε, μια πραγματική απαλωτρίωση. Κάποιοι χαμογελάνε με αυτά που λέω, αλλά έτσι είναι η κατάσταση. Μπορούμε να μιλάμε και για τις ε, τροποποίησεις οδηγιών, αλλά έχουμε και κάποιες κατευθύνσεις για την εφαρμογή των οδηγιών. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γιάλα Σέντερ. Ναι, ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι το πακέτο για την κυκλική οικονομία. Στην Ισπανία οι σοσιαλιστές ε, έχουμε προωθήσει αυτό τον κλάδο της επιλεκτικής προσέγγισης και έχουμε δημιουργήσει και μικρές αποκλειστικές αγορές. Είναι ένα πολύ σημαντικό πακέτο και σηματοδοτεί αλλαγή από τη μελέτη, την αρχή του πρώτου μέχρι την τελική ανακύκλωση και από τη πλευρά της βιομηχανίας αυτές οι αγορές, ε, οι μικρές αποκλειστικές αγορές είναι κάτι σημαντικό, πρέπει να το δημιουργήσουμε και συμφωνώ και σας συγχαίρω και πείτε μας πού μπορούμε να βοηθήσουμε, είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε γιατί έχουμε τεχνογνωσία. Θέλω επίσης να σας ενημερώσω για κάτι ακόμη. Σε σχέση με κάποιες ε, περιοχές όπου έχουν υπάρξει κάποιες ε, ε, διαθέσει αποβλήτων θα πρέπει να βρούμε κάποιες ε, λύσεις ε, βιομηχανικές. Δηλαδή δεν αρκεί να λέμε που βρίσκονται σοβαρά προβλήματα. Τα γνωρίζουμε αυτά τα προβλήματα και διονίζονται ορισμένα από αυτά. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε πλέον τεχνικές λύσεις όπως στην περίπτωση του Λιντέιν. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε και αν μπορείτε και εσείς να μας βοηθήσετε. Επίσης, εναγωνίως προσπαθούμε να νομοθετήσουμε. Είπατε κι εσείς, εφαρμογή είναι πρόβλημα. Μέσω κατεξοδότηση πράξεων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σας έχουμε βοηθήσει και, και εμείς από την πλευρά μας, σε αυτή την πολύ κρίσιμη στιγμή βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη νομοθεσίας για κάποιε περιπτώσει, Αναγνωρίζουμε όμω ότι το πρόβλημα δεν είναι να νομοθετεί κανεί, αλλά να εφαρμόζει τα νομοθετηθέντα. Και δεν ξέρω, μπορεί να είναι απαρχαιωμένη νομοθεσία, μπορεί να χρειάζεται αλλαγή ή όχι κτλ. Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή όμω, το Κοινοβούλιο δεν έχει το ρόλο που θα έπρεπε να είχε. Έχουμε τι κατεξουσιοδότε πράξει. Η Κομισιόν λοιπόν έχει αναλάβει το ρόλο για το τι γίνεται εκ των υστέρων. Επίση, Σημαντικό είναι να υπάρξει αυτή η σωστή εφαρμογή, αλλά τα κράτη-μέλη, κυβερνήσεις πρέπει να ε, κάνουν αυτό που πρέπει. Θα σας παρακαλούσα λοιπόν να, να έχουμε μια κοινή στάση και προσέγγιση, ανάλογα βέβαια με τους διάφορους κλάδους, αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσαμε σε αυτές τις κοινοβουλευτικέ συναντήσεις που έχουμε με τα εθνικά κοινοβούλια, που πολλές φορές ε, είναι πάρα πολύ επίσημες, τυπικές κτλ. Έρχονται οι βουλευτές, συναντούν και μιλούν ε, με τους ε, ομολόγους τους, αλλά δεν βγαίνει τίποτα από εκεί. Θα ήθελα να προσπαθήσουμε να δώσουμε στο κοινοβούλιο αυτό ένα σημαντικό ρόλο. Γιατί και εμείς μαζί με την Κομισιόν θα έπρεπε να ελέγχουμε αυτά που παράγουμε. Έχουμε την παραγωγή και τώρα ε, έχουμε την υλοποίηση. Κάπου εκεί μπορούσε να βρεθεί ο ρόλος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για να μην ζητάμε ή να απαιτούμε πράγματα τελικά που μπορεί και να αντιβαίνουν στη διάμεσα τα συμφέροντα. Μιλήσατε και για το ΕΦΣΙ, το Ταμείο Επενδύσεων. Εμείς προσπαθούμε με κάθε τρόπο να σας βοηθήσουμε. Σε κάποιες χώρες Το είχα πει και στον κύριο Κατάινεν στο Στρασβούργο στη συζήτηση που είχαμε υπάρχουν κάποιες χώρες που έχουν έλλειμμα εντό εισαγωγικών. Εκεί δεν μπορούμε να έχουμε ε, μια θετική εφαρμογή του λεγόμενου χρυσού κανόνα. Στο τι συνεισφέρει το κάθε κράτος ε, στον κοινό κορβανά δηλαδή. Τώρα έχουμε τις πλατφόρμες, τις τράπεζες ε, και εκεί έχουμε αντιμετωπίσει πραγματικά προβλήματα. Πώς θα βελτιώσουμε λοιπόν και τις δυνατότητες του ΕΦΣΙ αλλά και την αντίληψη που έχουν κυρίως οι δημόσιες δικής ορισμών κρατών μελών. Μπορεί να υπάρχουν χρήματα ε, στην τράπεζα, αλλά αφού αποφάσισε εμάς ο Υπουργός ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα, μπλοκάρισαν πολλά ε, προγράμματα. Μήπως μπορεί να βοηθήσετε λοιπόν τον Επιτρόπο Κατάινεν να προχωρήσει η εφαρμογή του χρυσού κανόνα σε άλλο επίπεδα, τοπικό, περιφερειακό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία ε, Κάντενβάχτε, τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Αντιπρόεδρε, ευχαριστούμε και για την υπομονή σα και ευχαριστούμε για την παρουσίαση που μα κάνατε. Αυτά που είπατε είναι σημαντικά. Το REFIT, η προσπάθεια για τη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου είναι σημαντικό για μα. Και αυτό που είπατε ότι αν κάτι δεν είναι χαλασμένο δεν χρειάζεται να κάνουμε προσπάθεια να το επισκευάσουμε. Αυτή είναι η θέση ε, την οποία θέλουμε να υποστηρίξουμε. Όταν λειτουργούν οι οδηγίε, δεν χρειάζεται να τι αλλάξουμε. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ασφάλεια δικαίου στα κράτη-μέλη και άλλοι συνάδελφοι το έθεσαν το όριο αυτό. Ε, μπορούμε να ακούσουμε από εσά πότε νομίζετε ότι θα υποβάλλετε ένα έγγραφο εργασίας με τις περαιτέρω δράσεις της Επιτροπής. Ε, δεύτερον, ε, Χάρηκα που άκουσα ότι είστε υπέρ της προστασίας της βιοπικιλότητας και θα περιμένουμε και εκεί τις ε, προτάσεις σας για να μπορέσουμε και εμείς ε, να βοηθήσουμε. Και μια ε, γενικότερη παράκληση προς εσάς για το ρόλο σας ως Αντιπροέδρου. Θα ήταν καλό να προωθήσετε την έκφραση της Επιτροπής με μία φωνή. Δηλαδή, όταν μιλάτε για την κυκλική οικονομία, καλό θα ήταν να υπάρχει μία κοινή πορεία όλων των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να συμβαδίζουν και με το άρθρο 168 όσον αφορά ε, τα θέματα υγείας, γιατί νομίζω ότι τα θέματα υγείας τα παραμελούμε λίγο αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους, λέει ο Πρόεδρος. Ε, πολλές ήταν οι ερωτήσεις. Και τώρα δίνω το λόγο σε εσά, κύριε Αντιπρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις και ζητώ εξ αρχής συγγνώμη αν μου διαφύγει κάποια ερώτηση. Θα προσπαθήσω να τις απαντήσω όλες. Κύριε Μπέλετ, σχετικά με ε, το ε, ερώτημά σας για τη σπατάλη των μέσων διατροφής. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε πολιτικές ώστε να παράγουμε λιγότερα απόβλητα και τα απόβλητα τα οποία υπάρχουν να τα χρησιμοποιούμε με τρόπο βιώσιμο και να μην θίγουμε το περιβάλλον. Φυσικά, εκείνο που θέλουμε να κάνουμε είναι να φροντίσουμε να μην υπάρχουν αυτές οι χωματερές. Αλλά από τη χώρα που γνωρίζω καλύτερα, γνωρίζω πολύ καλά ότι αν δεν προσέχει κανείς ε, μακροπρόθεσμα και κάνει βραχυπρόθεσμες επενδύσεις στις καύσεις, ε, τότε η δημιουργείται ζήτηση και το θέμα είναι πώς μπορεί κανείς με βιώσιμο τρόπο να λύσει αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό έχω ορισμένε αμφιβολίες. Πιστεύω ότι πρέπει να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη προκειμένου να αποκτήσουν μια ολιστική προσέγγιση που έχει σχέση με θέματα όπως το eco-design και άλλα, προκειμένου να μην υπάρχουν απόβλητα από την αρχή. Τώρα για την καύση. Η καύση των αποβλήτων είναι πολύ περίπλοκο θέμα. Διότι πρώτα απ' όλα λέμε δεν θέλουμε τους χιτά. Εντάξει, αυτό είναι σαφές. Υπάρχουν, υπάρχει αρκετή συμφωνία εδώ. Το επόμενο βήμα, κατά τη γνώμη μου, είναι πώς μπορούμε να περιορίσουμε την καύση στο ελάχιστο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει ποτέ κάψη ε, των αποβλήτων, διότι ακόμα και στην κυκλική οικονομία σε κάποιο στάδιο τα συστατικά που χρησιμοποιήθηκαν 4, 5, 6 φορές κάποια στιγμή φτάνουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους και ίσως η καύση να είναι απαραίτητη. Αλλά αυτό πάλι πρέπει να γίνει με βιώσιμο τρόπο. Έτσι θα έβλεπα το θέμα και νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε με τα κράτη-μέλη διότι όλοι δεν βρίσκονται στην ίδια φάση, στο ίδιο στάδιο σε αυτή τη συζήτηση. Υπάρχουν κρατημέλη που πάνω από το 50% ακόμα και περισσότερο χρησιμοποιούν χωματερές. Και ορισμενα κρατημέλη, ήμουν στην Εσθονία πριν από λίγο καιρό, από το 70% των χιτά σε λίγα χρόνια πέρασαν σε 9% νομίζω, σε πολύ χαμηλό ποσοστό χιτά. Συνεπώς είναι και θέμα ε, πολιτικών επιλογών και κινήτρων που υπάρχουν. Έχετε απολύτως δίκιο ότι το όλο θέμα είναι πώς μπορούν τα απόβλητα να είναι κάτι το επιθυμητό, να είναι αξιοποιήσιμα. Και σε πολλά κράτη-μέλη αυτό που βλέπω είναι ότι οι επιχειρηματίες ε, που ασχολούνται με τη διαχείριση των αποβλήτων, δεν μιλάω για βεντέτες, για σοπράνο, αλλά που με τη διαχείριση των αποβλήτων, σκέφτονται ποιο είναι το επιχειρησιακό μοντέλο, πώ μπορούν δηλαδή να κερδίζουν χρήματα από τα απόβλητα, εφόσον γνωρίζουν ε, ότι υπάρχουν και είναι αξιοποιήσιμα, προ το παρόν ξέρουν πώ να τα βάλουν στα χιτά ή στου καυστήρε. Αλλά παρακαλούμε, στρέφονται σε εμά και μα ζητούν να του προτείνουμε τρόπου ε, για να ανακυκλώσουν τα απόβλητα και να κερδίσουν χρήματα. Αυτή είναι πολύ καλή προσέγγιση προκειμένου τα άτομα που έχουν τη μεγάλη εμπειρία να τους βοηθήσουν και να μην τους λέμε απλά και μόνο ότι αυτά που κάνετε είναι λάθος και σταματήσετε, αλλά να τους βοηθήσουμε να κάνουν τη δική τους τη μετάβαση προς μια κατάσταση όπου χρησιμοποιούν τα απόβλητα με εποφελή τρόπο. Όπως είπαν μερικοί από εσά, το πρόβλημα εδώ είναι ότι χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση είναι το, ο σχεδιασμός, το design, η παραγωγή, οι πρώτες η ανακύκλωση. Για παράδειγμα, το τσιμέντο είναι το προϊόν το οποίο ρηπαίνει περισσότερο το περιβάλλον και χρησιμοποιείται σε τόσο ευρεία κλίμακα παγκοσμίω. Χρησιμοποιούμε περισσότερο τσιμέντο σήμερα σε ένα χρόνο από ό,τι χρησιμοποιούσαν ε, όλοι ε, στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία για να κτίσουν τα κτίρια τους. Και βλέπετε τι συμβαίνει σε πολλά μέρη του κόσμου. Αν μπορούμε λοιπόν να αλλάξουμε αυτό, δηλαδή ο οικοδομικός τομέας ε, να επαναχρησιμοποιεί το τσιμέντο και να βρεθούν και άλλες συναλλακτικέ λύσεις προς το τσιμέντο, τότε πραγματικά θα υπάρξει μείωση της ρήπανσης και αυτό θα σημαίνει πολύ μεγάλη πρόοδο στο, στην προστασία του περιβάλλοντος. Σημαντικό είναι να το γνωρίζουμε, αλλά πρέπει να ξανασκεφτείτε όλο τον οικοδομικό τομέα. Και νομίζω, τουλάχιστον για μένα, ότι αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, εάν μπορείτε να βοηθήσετε τις βιομηχανίες και τις χώρες να ακολουθήσουν τη σωστή κατεύθυνση. Λοιπόν, αυτό απαιτεί μια πραγματικά πολύ μεγάλη ολιστική προσέγγιση ε, και αυτό απαιτεί χρόνια δουλειά από μέρου μας. Στον κύριο Πόρσο, είμαι απόλυτα σαφής. Η Επιτροπή δεν έχει την πρόθεση να αποσύρει την οδηγία που αναφέρατε. Δεν είναι αυτή η πρόθεσή μας. Θέλω να είμαστε απόλυτα σαφείς εδώ. Για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες. Δεν θέλω να προδικάσω τα αποτελέσματα της συζήτησής σας που θα έχετε αύριο με τον κύριο Ανδριουκάκη Αλλά το θέμα είναι να ε, αναπτύξουμε τον ορισμό ε, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και να δούμε πώς μπορεί κανείς να εφαρμόσει σωστά και στην πράξη αυτόν τον ορισμό. Ε, συμφωνούμε απόλυτα με την ΠΟΗ και θα πρέπει για ορισμένους τομείς τα εντομοκτώνα, παρασυντοκτώνα, να γνωρίζουμε ποιες είναι οι νομικές μας υποχρεώσεις. Αυτές είναι οι μόνες λεπτομέρειες που μπορώ να σας δώσω αυτή τη στιγμή. Αν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειε προτείνω να έχετε σε επαφή με τον συναδελφό μου Άντριου Κάιτης. Τώρα, η δημόσια διαβούλευση. Το όνομά σας μου διαφεύγει, ζητώ συγγνώμη. Καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό που θέλετε να πείτε. Μερικές φορές και εγώ όταν άρχισα να με αυτό το μηχανισμό της δημόσιας διαβούλευσης, πω πω Θεέ μου, τα ίδια ακούμε, τα ίδια μηνύματα συνέχεια. Αλλά αργότερα, βλέποντα τα πράγματα από πιο κοντά, κατάλαβα ότι πολύ συχνά αυτοί οι άνθρωποι έχουν πάθος για αυτό το θέμα, αλλά δεν έχουν τα μέσα για να εκφράσουν με λόγια αυτό που σκέπτονται και τους βοηθούν άλλοι οι οποίοι διατυπώνουν τη δική του σκέψη και τελικά το μήνυμα που περνάει είναι το ίδιο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το άτομο που στέλνει το μήνυμα δεν εκφράζει τα πραγματικά του συναισθήματα και τις απόψεις του. Αν θέλετε λοιπόν μια δημόσια διαβούλευση, θα έχετε αυτή τη βοήθεια, διότι θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να οργανωθούν. Και ειλικρινά το ίδιο αισθανόμουν και εγώ στην αρχή. Σκεφτόμουν ότι ήταν αυτοματοποιημένες απαντήσεις. Πίσω από αυτό όμως υπάρχει ένα άτομο το οποίο συχνά αισθάνεται ότι πράγματι η απάντηση που δόθηκε ήταν εκείνη που θα έδινε ο ίδιος αν ήξερε να τη διατυπώσει. Λοιπόν, δεν απορρίπτω τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης επειδή ορισμένες απαντήσεις είναι πανομοιότυπες επειδή έχουν διατυπωθεί με τον ίδιο τρόπο. Βεβαίω δεν μπορώ να σας δώσω καμία εγγύηση ότι αυτό είναι αυτό που είπατε κι εσείς, αλλά προσωπικά εγώ έλεγξα αυτά που είπα, ρώτησα ορισμένου γιατί το είπαν και μερικές φορές το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο περίμεναν. Τελικά το αποτέλεσμα είναι ακριβώς αυτό το οποίο ήθελαν. Και γι' αυτό το λόγο είπαν ότι πιστεύω στη δουλειά που κάνει αυτή η οργάνωση και θέλω να την υποστηρίξω, θέλω η Επιτροπή και άλλοι να γνωρίζουν ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Νομίζω ότι αν εξυγχρονίσουμε τις δημοκρατίες μας, εάν, ας πούμε, ή, να δούμε τι υπάρχει γύρω μας. Οι Βρετανοί έχουν ταλέντα. Αν μπορούν λοιπόν να τα μεταφέρουν πατώντας ένα κουμπί, θα σκεφτούν επίσης πιο άμεσα τη δημοκρατία, εφόσον μπορούν να διατυπώσουν την άποψή τους πάνω σε θέματα που θεωρούν σημαντικά. Και όχι μόνο μέσω της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Δεν λέω ότι αυτή είναι μια εναλλακτική προ την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, αλλά ενισχύει τη δημοκρατία. Αν υπάρχει δημόσια διαβούλευση, α τη χρησιμοποιήσουμε ω σημαντικό μηχανισμό. Διότι με αυτόν τον τρόπο ο κόσμος μπορεί να διατυπώσει την άποψή του. Πιστεύω ότι αυτό ενισχύει τη δική σας τη δουλειά και τη δική μου τη δουλειά και δεν εξασθενίζει το έργο μα. Τώρα, για την επιτροπολογία. Αυτό το θέμα είναι πάντοτε ενδιαφέρον. Αφορά την πολιτική και τον τρόπο που λειτουργούμε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των συνθήκων. Έχουμε ορισμένα παραδείγματα. Ε, όταν ήμουν υπουργό, είχα ένα θέμα για τους ε, μη οργανισμούς. 28 χώρες. Τότε ήμασταν 26 χώρες που δεν ήθελαν αυτή την απόφαση. Αλλά επειδή ε, είχε τοποθετηθεί στην Επιτροπολογία, τίποτα δεν μπορούσαμε να κάνουμε, εκτός αν υπήρξαν επιστημονικά τεκμήρια προς το αντίθετο. Και υπήρχε ένας ανταγωνισμός, αν θέλετε, ανάμεσα στις πολιτικές επιλογές και στα επιστημονικά τεκμήρια. Και αυτό δεν είναι καλό. Είτε αποφασίζετε, εμείς αποφασίζουμε με βάση τα επιστημονικά τεκμήρια, πρέπει να δεχθεί κανεί αυτή την απόφαση και να ενεργήσει. Σχετικά ή λέτε ότι δεν το θέλουμε, θέλουμε να είναι πολιτική απόφαση και τότε πρέπει να αλλάξουν οι κανόνε και να γίνει πολιτική απόφαση. Τι συμβαίνει τώρα όμω. Και νομίζω ότι ο κ. Χάλτομα το είπε πάρα πολύ καλά. Τα κράτη-μέλη δεν ξέρουν πολύ καλά τι θέλουν να κάνουν, υπάρχουν εσωτερικές προστριβές. Το θέμα λοιπόν, το καλύτερο είναι η αποχή. Και η Επιτροπή δεν έχει την πολυτέλεια της αποχής, μερικές φορές θα ήθελε να απόσχει και θα έλεγε αν δεν θέλετε την πολιτική ευθύνη τότε μη μου την φέρετε στην πλάτη μου. Δυστυχώς δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Αλλά νομίζω ότι αργά ή γρήγορα και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας πρέπει να ξανασκεφτούμε κατά πόσον αυτό είναι ένας βιώσιμος τρόπος λήψης αποφάσεων. Δεν έχω απάντηση. Όπως κάνετε κι εσείς, απλώς επισημαίνω το πρόβλημα. Γιατί δεν έχω απάντηση, γιατί χρειαζόμαστε τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη πρέπει να δώσουν απάντηση. Αν θέλετε να μιλάμε μόνο σε πολιτικό επίπεδο, τότε λαμβάνετε η απόφαση στο Συμβούλιο. Αν όμως λέτε ότι θέλουμε ε, να, έχουμε ως βάση την επιστήμη και δεν θέλουμε παρεμβολή της πολιτικής, αλλά, και προσθέτω, προσέξτε, σε ποια θέματα θέλετε να έχετε επιστημονική βάση, διότι μπορεί να σας βαγκώσει εκεί που δεν θέλετε να σας βαγκώσει επιστήμη. Και αυτή είναι μια πρόκληση. Πάλι δεν έχω λύση να προτείνω. Αλλά απλώς και μόνο σας λέω το θέμα είναι πολύ λεπτό και θα πρέπει να το εξετάσουμε. Τώρα για τα εντομοκτώνα, γενικά παρασιτοκτώνα, μας ε, ενημερώς ε, αποφάσιστε ε, να παρακολουθεί το θέμα στην Επιτροπή Αναφορών στις 27 Ιουνίου. Θα εξακολουθούμε να βοηθούμε τα κράτη-μέλη για να βρουν μια λύση η οποία θα έχει την ευρύτερη δυνατή υποστήριξη και θα εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη προστασία τη ζωή και του περιβάλλοντο όπω προβλέπει η κοινωτική νομοθεσία. Πάντοτε με βάση τα επιστημονικά τεκμήρια που είναι διαθέσιμα. Αυτό είναι το τέλειο θέμα που βλέπετε ότι έχει πολιτικοποιηθεί τελικά. Τα επιστημονικά στοιχεία, πολύ καλά, ε, είναι καλά όταν είναι σύμφωνα με την πολιτική σας κρίση. Διαφορετικά είναι άχρηστα. Και αυτή είναι η κατάσταση όπου πιστεύω ε, δεν πρέπει να πέσουμε σε παγίδα. Τώρα, για τα απόβλητα τροφίμων. Τα εθνικά κοινοβούλια ε, το έθιξα το θέμα με την πρωτοβουλία για την πράσινη κάρτα. Και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό και πρέπει να καταλάβουμε πού χάνονται οι τροφές, πόσες τροφές χάνονται, γιατί χάνονται. Πώς θα υπάρξει διατροφή σε όλη την Ιφίλιο. Αν δούμε τη δημογραφική αύξηση δεν πρέπει να χάνονται τα τρόφιμα. Μιλάμε για τη διαχείριση των υδάτων, δύσκολη, δύσκολο θέμα. Ξέρετε όλα τα θέματα που πρέπει ε, να αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, χρειάζεται να έχουμε σωστή μέτρηση των επιπέδων τροφίμων που χάνονται στα κρατημέλη και επίσης ε, στην ε, αλυσίδα τροφίμων πώς μπορούμε να επεμβαίνουμε. Εδώ πρέπει και η βιομηχανία και τα κρατημέλη να συνεργαστούν όταν έχουμε μία πλατφόρμα όπου συμμετέχουν όλοι στην ε, ε, αλυσίδα τροφίμων, ώστε να υπάρχει μεταφορά πληροφοριών με βάση ε, στοιχεία απόλυτα σωστά. Πρέπει να υπάρχει συντονισμός με τις παγκόσμιες προσπάθειες που γίνονται και μπορείτε να βασιστείτε στη συνεχή υποστήριξη που θα σας παρέχω. Πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Πριν από το τέλος του χρόνου, σχεδιάζουμε να αναλάβουμε μια πρωτοβουλία για την πρόσφαση στη δικαιοσύνη. Ο δικό χάρτη θα δημοσιευτεί τι επόμενε ημέρε, που θα έχει τη μορφή ερμηνευτική οδηγία των αποφάσεων που έχει ήδη λάβει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όσον αφορά τη συμμόρφωση ε, επιθυμούμε να βελτιώσουμε τις μεθόδους που χρησιμοποιούν τα κρατη και να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση και επίσης εξετάζουμε αυτό το θέμα μαζί με τα κρατη εδώ και πολλά χρόνια στα πλαίσια της καλύτερης λειτουργίας και προσβλέπω στη συνεργασία σας αν έχετε σχόλια για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα. Παρακαλώ να μου τα στείλετε γραπτός με email. Θα σας ήμουν ευγνώμων. Όχι, δεν θα σας δώσω προθεσμίες. Αν θα σας δώσω προθεσμίες που είναι πολύ κοντές έχω πρόβλημα, αν θα σας δώσω πολύ μεγάλες προθεσμίες, τότε δεν θα κάνετε τίποτα, θα με μαλώσει η Κομισιόν. Δεν πρόκειται να έχετε προθεσμίες. Παρακαλώ δώστε μου λίγη ευελιξία. Εγώ θέλω να ενεργήσουμε γρήγορα, αλλά δεν δίνω προθεσμίες. Η ζωή μου θα γίνει πιο γρήγορη, πιο δύσκολη, γι' αυτό δεν πρόκειται να σας δώσω τις προθεσμίες. Είμαι βέβαιος θα μου δώσετε αποτελέσματα που περιμένω. Σε ό,τι αφορά τώρα... Α, όχι. Τι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε με τα πτηνά και τα οικοσυστήματα. Είναι το γεγονός ότι πολύ συχνά τα κράτη-μέλη ενώ έχουν κάνει αυτά λάθος, θα ρίχνουν αλλού. Δεν θέλω να είμαστε πάρα πολύ ευέλικτοι, να ανοίξω υπερβολικά τα περιθώρια, αλλά θέλουμε ευελιξία για να διευκρινίσουμε ποιος είναι υπεύθυνο γιατί. Διότι βαρέθηκα να κατηγορούνται οι Βρυξέλλες για τα λάθη που έκαναν οι χώρες μέλη με την νομοθεσία τους, την εθνική. Νομίζω ότι εδώ επιδέχεται το πράγμα βελτίωση. Για τον κύριο Παρνιό, για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, Υπάρχει κατάλογος ουσιών στην ε, ανάλυση αντικτύπου που δημοσιεύτηκε σήμερα και σας παραπέμπω στον κατάλογο αυτό. Πρόκειται για μία μελέτη και όχι για επίσημο έγγραφο και γι' αυτό ζητήσαμε από την ΕΦΣΑ, την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, να κάνει ένα screening, όπως λέμε στα γαλλικά, για τις ουσίες που θα μπορούσαν να είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες Ε, διαφάνεια και καπνός. Εδώ δεν συμφωνώ με την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, διότι η προσέγγιση μας είναι γνωστή σε ό,τι αφορά τους γενικούς διευθυντές, τα μέλη πολιτικών γραφείων κτλ. Η γάμα δέλτα υγεία, νομίζω, σαν τε, υιοθέτησε μονομερός μια θέση. Τώρα μας λέει η διαμεσολαβήτρια, αυτή την προσέγγιση της μίας γενικής διευθύνσης πρέπει να την διευρύνεται να την επεκτείνει σε όλες τις άλλες. Ήρθα σε επαφή με την διαμεσολαβητρία και αναλύσαμε το κατά πόσον αυτό είναι αναγκαίο ή συνιστά πολύ μεγάλο φορτίο λόγω των αποτελεσμάτων. Επειδή τώρα έχουμε την νομοθεσία σε ίσχυ ε, και επειδή οι επαφέ μα με την καπνοβιομηχανία είναι πάρα πολύ περιορισμένε, ιδίω για τι άλλε γαμαδέλτα, θα ήταν υπερβολή να επιβάλλουμε το ίδιο καθεστώ σε όλη την Κομισιόν. Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσα λοιπόν στην άποψη τη Διαμεσολαβήτριας. Για τους ανθρωπινικούς διδάκτες τα είπα, για τα τρόφιμα, για τα απόκτα τα είπα, για τους νέους. Ναι, εδώ θέλω να επιμείνω. Το ΕΦΣΙ, αυτό το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, επιτυγχάνει στις χώρες εκείνες όπου η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τοπικές τράπεζες ε, τοπικές τράπεζες επενδύσεων και οργανώσεις επιχειρηματιών διασυνδέονται μεταξύ τους. Τότε έχουμε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο μόχλευσης. Ένα στα 15 νομίζαμε είναι ένα στα 23. 23 φορές παραπάνω. 23 ε, ε, φορές παραπάνω είναι μεγάλο πράγμα. Και είδα πολλοί νέου επιχειρηματίε από την Ολλανδία χθε, οι οποίοι μέσω του ΕΦΡΟ και του ΕΦΣΙ, αλλά στρέφονται τώρα και στο ΕΦΣΙ, και βλέπουν ότι είναι τεράστια αυτή η ευκαιρία, γιατί οι επενδύσεις συνήθω πηγαίνουν ε, στι μεγάλε βιομηχανίε. Ε, τώρα βλέπουμε αλλαγή με το ΕΦΣΙ και το μέλλον είναι στι μικρομεσαίε επιχειρήσει, αν δείτε. Όλα ό,τι έχουν να κάνουν τι ανανεώσιμες πηγέ ενέργεια, την αλλαγή νοοτροπία, για την στέγαση, την κατοικία. Όχι, δεν μιλάμε πλέον για κατανάλωση, αλλά για παραγωγή ενέργεια κτλ. κτλ. Τεράστιες αλλαγές. Χρειαζόμαστε ΜΜΕ. Για να στεφθεί με επιτυχία αυτή η προσπάθεια, ε, οι νεαροί επιχειρηματίε, οι νοφεί επιχειρήσει είναι αυτέ που θα πρέπει να διασνεθούν σε αυτή την προσπάθεια και αυτό αναζητεί και ο Κάρλο Μοέδα. Για την υγεία τώρα. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι μας διέ... γνώμονας είναι οι πολιτικές για την υγεία και θέλουμε να έχουμε βιώσιμα συστήματα υγείας. Και επειδή μιλάω για βιωσιμότητα. Ο κόσμος γιατί ανησυχεί γιατί φοβάται ότι η πρόσβαση στις ε, θεραπείες, ε, στους γιατρούς ε, θα περιοριστεί λόγω των πληθυσμιακών αλλαγών, δημογραφικής ανάπτυξης κτλ. Αν θέλουμε λοιπόν τα συστήματα, τα κοινωνικά και τα συστήματα υγείας να εξακολουθήσουν να παρέχουν υπηρεσίες, θα πρέπει να μας απασχολήσει η βιωσιμότητα μακροπρόθεσμα. Και νομίζω ότι έτσι θέλουν να ζουν οι Ευρωπαίοι. Και σίγουρα προσπαθήσουμε και εμείς από το δικό μας μετερίζει να το υποστηρίξουμε για το ΕΦΣΥ. Μίλησα για την κυκλική οικονομία. Μίλησα να επιβεβαιώσω και προς την κυρία Κάντεμπαχ ότι δεν θα σας δώσω σήμερα προθεσμία. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας ε, και λυπούμε που μακρηγόρησα πάντα σε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα και γιατί το γεγονός ότι απαντήσατε σε όλες μας ερωτήσεις. Νομίζω τώρα ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες σας και θα σας δούμε αύριο το πρωί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και ιδίω ευχαριστώ τον κύριο Τίμερμαν, τον κύριο Αντιπρόεδρο, για την παρουσία του και για το γεγονός ότι απήντησε σε όλες μας τις ερωτήσεις.